Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ήθελα απλώς να πω ότι ψήφισα υπέρ, αλλά η κονσόλα δεν λειτουργούσε. Θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά, κυρία Κορόλα. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους καλή επιστροφή στα σπίτια τους στην περίπτωση που ε, λόγω δυσχερών κλιματικών συνθήκων ή απεργία στη Γερμανία ε, δυσκολευτούν να πάνε στο σπίτι τους. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι στη Γερμανία την πέμπτη, σήμερα την Πέμπτη ε, υπάρχει το, το, συνήθιο να κόβουν τις γραβάτες των ανδρών στο πλαίσιο του καρναβαλιού. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί με τις γραβάτες σας.